La seduta Ξεκινάει η συνεδρίαση. Πριν λοιπόν περάσουμε στο σημείο της μήνυσης διάταξης που αφορά τις δηλώσεις του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα και επ' αυτού του θέματος ε, έχουν κατεκτεθεί 1224 τροπολογίες. Είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες και πολλές έχουν ζητηθεί να ψηφιστούν και χωριστά σε τμήματα. Ε, έχοντας λοιπόν συζητήσει με την Επιτροπή Μεταφορών, αποφάσισε να εφαρμόσω το άρθρο 165 του κανονισμού και να μεταθέσω, να αναβληθεί αυτό το θέμα και να υπάρξει πριν από την επόμενη ψηφορία η απαραίτητη προκαταρκτική εργασία, η προετοιμασία δηλαδή. Και έτσι, αποφάσισα να μπορούμε όταν πια θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε κανονικά με απόλυτη σαφήνεια. Είναι μια απόφαση την οποία έλαβα λαμβάνοντας υπόψη όλες ε, τις ε, απαραίτητες παραμέτρους ε, για να μπορούμε να έχουμε και μια σωστή αντιμετώπιση των τροπολογιών αλλά και να διασφαλίσουμε μια σαφή ψηφοφορία για τα βασικά θέματα. Αποφάσισα λοιπόν, σεβόμενος ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου, που πιστεύω ότι τα μέλη δεν μπορούν να αναγκαστούν να κάθονται όλες αυτές τις ώρες για να ψηφίζουν, κυρίως για τροπολογίες που δεν είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν και τροπολογίες που αν πρέπει να κρίνω από αυτό που έγινε τη Δευτέρα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο λάθους, μάλιστα υψηλότατο περιθώριο λάθους. Και έτσι, βάσει τον κανονισμό 206 του κανονισμού υπαριθμών 1, καλώ την Επιτροπή Μεταφορών να συνέλθει ε, την Δευτέρα και την Τρίτη έκτακτα και να υποβάλει στην Ολομέλεια το αποτέλεσμα των εργασιών της ε, και μάλιστα σε κατάλληλο χρόνο για να μπορούμε να ψηφίσουμε στην επόμενη ε, Ολομέλεια που θα είναι την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 165 του κανονισμού, οι τροπολογίες ε, που έχουν ζητηθεί, που θα κατατεθούν και εκείνες οι τροπολογίες που θα ψηφιστούν χωριστά και δεν θα εγκριθούν τουλάχιστον από το 1 τρίτο των μελών της Επιτροπής, αυτές δεν θα κατατεθούν στην Ολομέλεια. Και επιπλέον δεν θα είναι δυνατόν να κατατεθούν και άλλες ε, τροπολογίες ε, που θα ζητηθεί που θα πρέπει να ψηφιστούν σε χωριστά τμήματα. Είμαι λοιπόν <clears throat> σίγουρος ότι η Επιτροπή Μεταφορών θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και θα ήθελα να ενημερώσω την Ολομέλεια ότι έχοντας κατά νου αυτήν την απόφαση που έλαβα να ε, αναβάλουμε την ψηφορία για να λυθεί το θέμα των τροπολογιών, αυτό που ε, ζήτησαν ε, ε, πολλοί ευρωβουλευτές με βάση το άρθρο 185, αυτό το αίτημα κατέπεσε. Και όσον αφορά τη συζήτηση, οι συζητήσεις θα γίνουν όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Ερντογκ. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, είναι δικαίωμα σας να λάβετε την απόφαση αυτή, τη σέβομαι, αλλά ο κανόνας 175 προβλέπει επίσης ότι στην Επιτροπή με το 1 τρίτο των μελών της Επιτροπής μπορεί να αποφασιστεί αν οι τροπολογίες θα ε, ε, δοθούν πάλι στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα γίνει. Οπότε σε μια εβδομάδα θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όπως σήμερα. Το πρόβλημα δηλαδή δεν θα λυθεί από την Επιτροπή Μεταφορών όπως προβλέπετε. Υπάρχει αυτή η αναβολή κατά μία εβδομάδα, το θέμα θα παραμείνει ως έχει. Αγαπητέ, ε, προβλέπετε στον κανονισμό και διαβουλεύτηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, την πρόεδρο, και μου είπε ότι πράγματι ε, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ε, αυτό το αίτημα, αυτό που της αναθέσαμε. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τεχνικό αυτό το ζήτημα. Το άρθρο 175 αφορά τα κείμενα που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή. Πώς έχει η νομική κατάσταση τώρα. Γιατί έχουμε το θέμα της απόσπασης και το θέμα αυτό δεν προήλθε από την Επιτροπή, αλλά από πολλούς και διάφορους τρόπους. Τι ισχύει τελικά από τον εσωτερικό κανονισμό, ε, ποια άρθρα πρέπει να εφαρμοστούν, τι προβλέπετε. Chiudiamo il dibattito perché non dobbiamo aprire un dibattito su questo. Α κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, δεν πρέπει να ξεκινούμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ήθελα και σα ενημέρωσα για την απόφαση που ελήφθη με βάση τον κανονισμό και την απόφαση την έλαβα αφού διαβουλεύτηκα με την πρόεδρο τη Επιτροπής Μεταφορών. Το πρόβλημα είναι, όπω σα είπα, ο τεράστιο αριθμό των τροπολογιών και ο τεράστιο αριθμό τροπολογιών που ζητήθηκε να ψηφιστούν σε χωριστά τμήματα. Εάν τώρα υπάρχουν κάτι κάποια θέματα που πιστεύετε ότι είναι στοιχεία κολυσιεργίας. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά ισχύει και το άλλο, ότι ένα τμήμα, ένα κομμάτι αυτών των τροπολογιών ε, είναι, έχουν πολύ σημαντικό αντικείμενο. Άρα δεν πρόκειται για κολυσιεργία, αλλά πρόκειται ε, για ουσιαστική προσπάθεια να υπάρξουν παρεμβάσει στο κείμενο. Επειδή λοιπόν ε, το θέμα είναι πολύ περίπλοκο, δεν είναι ότι μπορούμε να ψηφίσουμε 4.000 φορές για ένα θέμα, εγώ σκέφτηκα να απευθυνθώ στην Επιτροπή Μεταφορών και την επόμενη εβδομάδα, εντάξει, αν δεν υπάρξει λύση, ας ψηφίσουμε για όλες τις τροπολογίε. Εγώ προσπάθησα να πείσω τους βουλευτές ε, ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ε, είδατε τι έγινε προχθές. Ε, εάν έχουμε τώρα 3.000 τροπολογίε στην Ολομέλεια, θα γίνει, θα ψηφίζουμε πράγματα που κανεί δεν καταλαβαίνει τι είναι προσπάθησα να πω συγκεντρώστε τις πληροφορίες. Το ECR είπε ότι είναι κατά αυτή τη ε, συγκέντρωση και του συνδυασμού των τροπολογιών και θέλει ε, ξεχωριστές ε, τροπολογίες. Ε, τώρα δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί κανεί να κάνει και να είναι σωστό για την τροπολογία. Α πούμε, κλείσουμε λοιπόν, ε, η Επιτροπή Μεταφορών θα κάνει τη δουλειά τη και θα δούμε στην επόμενη Ολομέλεια, στι Βρυξέλλες, θα δούμε τότε αν θα πρέπει να ψηφίσουμε 6.000 φορέ, α ψηφίσουμε 6.000 φορέ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Απλά ήθελα να κάνω μια προσπάθεια για να αντιμετωπίζονται οι βουλευτέ με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Η πρόεδρο τη Επιτροπής Μεταφορών με διαβεβαίωσε ότι μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά και γι' αυτό ας ε, ψηφίσουμε τότε πια το τι θα μας έχει παρουσιάσει η Επιτροπή Μεταφορών. Αν τώρα η Επιτροπή Μεταφορών μας καταθέσει 6.000 τροπολογίες, θα ψηφίσουμε για τις 6.000 τροπολογίες. Τώρα έκλεισε το θέμα. Κλείνει το θέμα κλείνει και περνάμε στο θέμα που είναι ε, συζήτηση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου, συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. δήλωση τη Επιτροπής για τα συμπεράσματα τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 21 η 22 η ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τούσκα και από τον κύριο Γιούνκα για αυτή την καθυστέρηση, αλλά όπως ξέρετε και εσείς, ε, η δέσμη μέτρων για την κινητικότητα έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις, διχασμό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι και προς όφελος του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώσω τους βουλευτές για την απόφαση μου. Κύριε Τούσκ, έχετε το λόγο ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη στο φως του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι ε, μια αυξημένη ταχύτητα στον τομέα αυτό θα αυξήσει την ευημερία αλλά και το ρόλο μας στην παγκόσμια σκηνή. Έτσι λοιπόν ελάβαμε έναν αριθμό πρωτοβουλειών. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να εμβαθυνθεί και να ενισχυθεί περισσότερο με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία την ψηφιακή και την οικονομία των υπηρεσιών. Ε, φραγμοί αδικαιολόγητοι πρέπει να απαλληφθούν, νέοι δεν πρέπει να δημιουργηθούν. Η Κομισιόν εκλήθη μέχρι το Μάρτιο του 2020 να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης μακροπρόθεσμο για καλύτερη εφαρμογή ε, και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Δεύτερον, συζητήσαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεδομένης της σημασίας της για εκατομμύρια θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, η Κομισιόν εκλήθη να παρουσιάσει ένα όραμα για το βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης ε, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο την ψηφιακή οικονομία της με ιδιαίτερη εστίαση στην, ε, στα δεδομένα και στην ε, τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίξαμε μια σύντονη προσέγγιση ε, με ενίσχυση των δικτύων 5G. Η Κομισιόν υπέβαλε σύσταση στον τομέα αυτών. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, το εμπόριο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να προάγει ε, ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που βασίζονται στο ε, ισότιμο ανταγωνισμό. Ε, το μηχανισμός των δημοσίων συμβάσεων συζητήθηκε από τους ηγέτες και η ταχεία εφαρμογή όλων των στοιχείων της κοινή δήλωσης της 25ης Ιουλίου του 2018 μεταξύ Ένωσης και ΕΠΑ. ΕΕ. Συζητήσαμε επίσης τις οικονομικές μας σχέσεις με την Κίνα. Εκτός ε, από το Σύνοδο Κορυφής ε, τον επόμενο μήνα Ένωση Κίνας υπάρχουν και άλλες συναντήσεις και σύνοδοι με τους Κινέζους ηγέτες. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε για μια, ε, επί μια συντονισμένης προσέγγισης. Είναι φιλόδοξη συνεργασία σε παγκόσμια θέματα συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου. Ε, έχουμε ένα κέριο οικονομικό συμφέρον και οι δύο στη διατήρηση νόμων του εμπορίου που στηρίζονται σε ένα σύστημα εμπορίου βασισμένου σε κανόνες. Για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα όμως θα πρέπει να εξυγχρονιστεί τάχιστα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ που θα καλύπτει τις βιομηχανικές επιδοτήσεις ως προτεραιότητα. Επίσης, πρέπει να πείσουμε την Κίνα να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και είμαι πεπισμένος ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, να παρατηθούμε. Εις ό,τι αφορά τα διμερή θέματα, θέλουμε να οριστικοποιήσουμε την Συμφωνία Επενδύσεων ήδη του χρόνου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Κίνα στην επικείμενη σύνοδο. Και βέβαια δεν φαντάζομαι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι το ίδιο σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το εμπόριο. Επίσης, ε, οι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Παρά τις διαφορές, είναι σαφές πόσο κατεπήγον είναι το θέμα. Οι ηγέτες θα επανέλθουν στο θέμα τον Ιούνιο. Στο ενδιάμεσο έχουμε δώσει οδηγίες στους υπουργούς να συνεχίσουν με περισσότερη προσπάθεια την μακροπρόθεσμη στρατηγική για να υλοποιηθούν οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων. Περνώ στο Brexit. Όπως ζήτησε η Πρωθυπουργό Μέη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη λεγόμενη Συμφωνία του Στρασβούργου. Οι ηγέτες επίσης εξέτασαν το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για σύντομη παράτηση της περίοδου βάσει του άρθρου 50. Η απόφασή μας για την παράταση προβλέπει δύο σενάρια. Πρώτον, αν η συμφωνία περάσει αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή των Κοινοτήτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί για μια τεχνική παράταση μέχρι τις 22 Μαΐου. Δεύτερον, στην περίπτωση που δεν θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων αυτή την εβδομάδα η συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε μια παράταση μέχρι τη 12η Απριλίου, περιμένοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο να υποδείξει την μελλοντική πορεία. Όπως είπα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί κέρια ημερομηνία τη 12η Απριλίου για να αποφασίσει το ε, Ηνωμένο Βασίλειο αν θα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Η 12η Απριλίου ε, είναι ε, ένα ορόσημο. Πριν από αυτή την ημερομηνία, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να διαλέξει συμφωνία, μη συμφωνία, μακρά παράταση ή ανάκληση του άρθρου 50. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια προσωπική παρατήρηση προς τα μέλη του Κοινοβουλίου. Πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπα ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε μια μακρά παράταση αν θέλει να επανεξετάσει το Ηνωμένο Βασίλειο τη στρατηγική του Brexit. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει στις ευρωεκλογέ. Και μετά ακούστηκαν φωνές που έλεγαν ότι αυτό θα είναι επιζήμιο ή μη εξυπηρετικό για πολλούς από εσά. Να ξεκαθαρίσω, μια τέτοια, ένα τέτοιο σκεπτικό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί τα 6 εκατομμύρια να τα γνωρίσουμε που υπέγραψαν την ανάκληση του άρθρου 50 τους ανθρώπους που ζήτησαν ε, νέα ψήφο ή τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που ζήτησαν παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορεί να θεωρήσουν ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να νιώθουν ότι εκπροσωπούνται σωστά από εσά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι Ευρωπαίοι. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιούγκερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Έχουμε ενώπιον μας μία εβδομάδα πλούσια σε εξελίξεις και γεγονότα. Κάτι που δεν με θαρρύνει να σχολιάσω και τα υπόλοιπα γεγονότα που έχουμε μπροστά μας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχαμε μια πολύ έντονη εβδομάδα, πολύ σημαντικές εξελίξεις και πολύ κομψά παρουσίασε τα διαμηθέντα στο Συμβούλιο ο Πρόεδρος Τούσκ. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που είπε. Συζητήσαμε εκτενώς το θέμα της Κίνας. Η συζήτηση για την Κίνα βέβαια ήταν λιγότερο περίπλοκη από τη συζήτηση για τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Έλεγα σε κάποιους από εσά ότι αν συνέκρινα την ε, Μεγάλη Βρετανία με τη Σφίγγα, η Σφίγγα μου φαίνεται ανοιχτό βιβλίο σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Και δεν ξέρω πότε επιτέλους το κλειστό βιβλίο της Μεγάλης Βρετανίας θα ανοίξει για να μιλήσει. Θα δούμε, ίσως χρειάζεται κατάλληλη στιγμή. Μιλήσαμε για την Κίνα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στις 12 Μαρτίου υπέβαλε την ε, στρατηγική της και ήταν πολύ θετική υποδοχή αυτού του εγγράφου. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων μίλησαν για τις αδρές γραμμές της κινέζικης στρατηγικής, κάτι που υποβάλαμε για διαλογισμό στο Συμβούλιο. Και μάλιστα με πρόταση του Πρόεδρου Μακρό θα δούμε και σε συνεργασία με την κυρία Μέρκελ θα συναντήσουμε τον Πρόεδρο ε, της Κίνας και ε, ήμασταν ε, σαφέστατοι ότι ως προς την Κίνα θα πρέπει όλοι να καταλάβουν και στην Ευρώπη και στην Κίνα ότι είμαστε εταίροι, στρατηγικοί εταίροι. Είμαστε ταυτόχρονα όμως και ανταγωνιστές και αντίζηλοι, αντίπαλοι. Διαπίστωσα σε κάποιες επαφές και συνεδριάσεις ότι οι Κινέζοι φίλοι μας ε, βλέπουν κάπως αρνητικά την έννοια του αντίπαλου του αντίζηλου. Αυτό όμως είναι κοπλιμέντο, φιλοφρόνηση. Σημαίνει ότι είμαστε ε, ανταγωνιστές, ισότιμοι και δεν θέλουμε να, να αυτοπαρουσιαστούμε ως Ευρώπη κλειστή, αλλά ανοιχτή. Ούτε φυσικά θα είμαστε ξέφραγο αμπέλη. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ε, και να τους εξασφαλίσουμε ανταγωνισμό σε κανονικούς όρους στην Κίνα. Το ίδιο και για τις κινέζικες επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμούς. Και σεβόμαστε την Κίνα, αλλά φυσικά θα θέλαμε να μας σεβαστεί και η Κίνα. Οπότε η εμπορική μας προσέγγιση χαρακτηρίζεται από μια απόλυτη αμοιβαιότητα απαιτούμε φυσικά να συμφωνήσουμε και εμείς ως προς μια συμφωνία για τις επενδύσεις και, ε, και η Κίνα θα πρέπει να δεχθεί την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και θα θέλαμε η ομάδα εργασίας που συστήθηκε με συμμετοχή Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αυτή η ομάδα εργασίας να προχωρήσει με κάποια ταχύτητα. Ίσως όχι ολικιώδη, αλλά με κάποια ταχύτητα. Για τον Brexit δεν θα πω τίποτα, γιατί ό,τι ήταν υποθεί, υπόθηκε. Merci, Monsieur le Président de la Commission européenne. timing. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τηρήσατε και το χρόνο σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Μάνφρεντ Μπέμπερ. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την καλή απόφαση για το Brexit, κύριε Τούσκ Νομίζω ότι η απόφαση του Συμβουλίου ήταν μια πολύ καλή απόφαση. Πρώτα απ' όλα διότι ε, συμπεριλήφθηκε και η αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρξει παράταση χωρί ε, διευκρίνηση από πλευρά ε, των Βρετανών φίλων μα για το τι ακριβώ επιθυμούν. Επίση, αυτό δημιουργεί κάποια ασφάλεια για, τους, για τα 400 περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίων σχετικά με τι ευρωεκλογέ. Αναφέρομαι στην ουσιαστική και την νομική ασφάλεια. Θα πω λιγάκι για αυτού αυτούς που αναφέρετε κι εσείς, ε, αυτούς που θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε μαζί τους, ε, τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία, αλλά προς το παρόν υπάρχει η κατάσταση και η απόφαση, η νομική απόφαση ότι η Μεγάλη Βρετανία θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας αυτό κατά νου, νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στους πολίτες μας γιατί μια χώρα που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή να πρέπει να της επιτραπεί να έχει λέγει στο τι θα γίνει στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα που θέτουν οι πολίτες και εκεί το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει ε, διευκρίνηση της κατάστασης και όχι ε, παράταση ε, εν λευκό. Θα ήθελα να ευχηθώ στους συναδέλφους μας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο να τα καταφέρουν καλύτερα. Έχουν πάρα πολλές επιλογές, είναι σαφείς αυτές και τώρα πλέον πρέπει να διαλέξουν. Ας δούμε τι θα κάνουν. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω έχει σχέση με την οικονομία και θέλω να σας πω ότι εμείς στηρίζουμε απολύτως τις αρχές περί ενίσχυσης της οικονομίας επενδύσεις στην κοινή αγορά, στην ε, καινοτομία, καμία αμφιβολία από αυτού. Βεβαίως προτεραιότητα είναι ε, το θέμα της Κίνας. Έχει τεθεί, ε, συζητιέται και είμαι ευγνώμων που όλοι συμμεριζόμαστε το ίδιο σημείο κίνησης. Δηλαδή η συνεργασία με την Κίνα πρέπει να βασίζεται σε αρχές. Συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για τα πολιτικά συστήματα συστήματα για το πώς ε, ε, οργανώνουμε μια κοινωνία, ποιες είναι οι βασικές αξίες μιας κοινωνίας και θεωρώ ότι αυτό πρέπει πάντα να είναι η αφετηρία για τι σχέσει μα με την Κίνα. Ω ΕΛΚΑ θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια ρεαλιστική προσέγγιση Ω προ την κλιματική αλλαγή. Η Κίνα εξακολουθεί να είναι δεσμευμένη με τη Συμφωνία των Παρισίων στο ελεύθερο εμπόριο και εκεί έχουμε σχέσει με την Κίνα. Έχουν δεσμευτεί οι Κινέζοι για το ελεύθερο εμπόριο. Άρα δηλαδή έχουμε την ίδια ρεαλιστική προσέγγιση. Το τρίτο όμω είναι εξίσου σημαντικό ότι δεν πρέπει να είμαστε αφελεί. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε τη δική μα μας βιομηχανία, την βασική βιομηχανία, ε, να την προστατεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς επίσης ως ΕΛΚΑ θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και θέματα ανταγωνισμού έτσι ώστε στο μέλλον να γίνουμε πρωτοπόροι και να μπορέσουμε να προσαρμέσουμε τη διάσταση του ανταγωνισμού ε, στα δικά μας τα θέματα. Θα ήθελα να δείξω και ένα τελευταίο θέμα, δηλαδή το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Τούσκα, εδώ και κάποιους μήνες ε, Έχουμε το θέμα του άρθρου 7 με την Πολωνία και την Ουγγαρία. Το Κοινοβούλιο το έθιξε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέχρι τώρα στο Συμβουλίο δεν υπήρξε καμία ευκαιρία να γίνει συζήτηση από αυτού. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το δικό μου το κόμμα, ε, φαντάζομαι θα το έχετε καταλάβει πολύ, είχε μία έντονη συζήτηση επί του θέματο. Αποφασίσαμε το ΦΙΝΤΕΣ, το Ουγγρικό ε, Κυβερνών Κόμμα, να ανασταλεί η συμμετοχή του στο ΕΛΚ, να μην έχει βασικά δικαιώματα. Άρα δηλαδή αυτό είναι ένα μήνυμα που εκπέμπουμε στην Ουγγαρία. Έχουμε το άρθρο 7 εντό στο Κοινοβούλιο που το στηρίξαμε ανεπιφύλακτα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πολύ επιτέλους να συζητήσετε για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τον επιτίθεται το ένα στον άλλον δημόσια. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά είναι ένα τελείω διαφορετικό θέμα να γίνονται ουσιαστικέ σοβαρέ εσωτερικέ συζητήσει. Να προσπαθήσετε κι εσεί. Όπω προσπαθούμε κι εμεί να συζητάμε με του Ρουμάνου φίλου, με το ΕΛΚ και με άλλου. Αυτό είναι ο σωστό τρόπο, να συζητάει κανεί και να λαμβάνει και αποφάσει. Επιθυμώ επίση να κάνουμε και ένα βήμα περαιτέρω. Δηλαδή, ε, το άρθρο σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να οδηγήσει ταχύτατα στα ευκταία αποτελέσματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι ένας ε, δεσμευτικός μηχανισμός ε, κράτους δικαίου που θα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επ' αυτού δούλεψαν πάρα πολλοί συνάδελφοι να έχουμε λοιπόν αυτό τον δεσμευτικό μηχανισμό ο οποίος θα διασφαλίζει ότι κάθε χρόνο θα υποβάλλεται μία έκθεση και θα ελέγχονται όχι μόνο οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά το σύνολο των κρατών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ελέγχονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε αυτές τις χώρες. Ε, επίσης, ε, δεν ξέρω τι θα γίνει με αποκλήσεις που ενδεχομένω μπορεί κανείς να ε, ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ ε, συνδέονται βέβαια και τα κονδύλια τα οποία διατίθενται. μπορούμε να είμαστε πιστικοί στη συζήτηση με την Κίνα ως ε, προς ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, μόνο αν και εμείς αυτές τις αξίες τις εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, κύριε Τούσκ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω επιτέλους το θέμα αυτό να το θέσετε στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δηλαδή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γίνουν συζητήσεις για τα θέματα που έχουν τεθεί επιτάπητο στην Ευρώπη. Το λόγο έχει ο κύριος Μπούλμαν εκ μέρους των σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε ακόμα δύο μέρες που απομένουν μέχρι την αρχική πρόβλεψη αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύο μέρες μένουν. Πρόεδρε Τούσκ, σωστό ήταν αυτό που προέβλεψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για να αποφύγει τα χειρότερα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι δύο μέρες πριν από την αρχικά προβλεφθή σε ημερομηνία εξόδου και απευθύνομαι στους υπέρμαχους του Brexit. Πότε θα έχετε την εντιμότητα να, να ζητήσετε συγνώμη από τον Βρετανικό λαό για τη στάση σας. Να έχετε την εντιμότητα να παραδεχτείτε ότι δεν ξέρατε τι κάνατε και δημιουργήσατε μια κατάσταση με υπενιγμούς από την οποία δεν γνωρίζατε πώς θα βγείτε. 10% ε, μειώθηκε το ΑΕΠ και εσείς δεν ξέρετε πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ε, πραγματικά πρέπει να παραδεχτείτε τα λάθη σας, τις υποκρισίες σας και να ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό είναι το βασικό μου μήνυμα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Τούσκ, για όσα κάνατε για να προασπίσετε την ευρωπαϊκή ε, ταυτότητα και ηθαγένεια. Είμαστε Ευρωπαίοι και κανείς δεν επιτρέπεται να εξαπατά το Βρετανικό λαό ε, και να του στερεί τη δυνατότητά του να συνεχίζει να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά πράγματα στο βαθμό που δεν προβλέπεται έξοδος. Ε, η κατάσταση αυτή παραμένει αποκλεισμένη και το μόνο που μένει να γίνει και το μόνο σωστό είναι να ερωτηθεί ο Βρετανικός λαός. Δεν θέλετε να το κάνετε γιατί φοβάστε, φοβάστε γιατί δεν τους επηρεάζετε πια. Αυτό θα ήταν η λύση και ο Βρετανικός λαός θα σας υποδείξει που προς τα που θα κινηθείτε γιατί είναι ο μόνος κυρίαρχος εν προκειμένου. Να πω επίσης ότι πιστεύω ότι βέβαια οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο επισκιάζει πολλά από αυτά που πρέπει να ρυθμίσουμε κατεπηγόντως. Στις 9 Μαΐου το επόμενο Συμβούλιο πρέπει να ασχοληθεί με μια μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την αναζωγόνηση της οικονομίας. Θέλουμε μια βιώσιμη οικονομία η οποία θα φίδεται του πλανήτη μας, ε, δεν θα κατασπαταλά τους πόρους και θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες συμμετοχή σε όλους. Αυτό πρέπει να είναι το θεματολόγιό μας. Και μόνο αν εμείς είμαστε ισχυροί, με αυτοπεποίθηση, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της Κίνας. Ρεαλιστικά βλέπουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν ισχυρότατο εταίρο που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Πρέπει όμως να έχουμε αυτοπεποίθηση, πρέπει να γνωρίζουμε τη δική μας θέση και δράση. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προασπίσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο. Εκεί θα συνεργαστούμε και ε, προς αυτό είναι πρόθυμη η δική μου ομάδα. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των ε, συντηρητικών μεταρρυθμιστών το λόγο έχει ο κύριος Λεγκούτκο, ο πρόεδρος της ομάδας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Πάντα έχουμε και χαρμόσυνες ειδήσει και κακά μαντάτα. Το καλό είναι ότι το Συμβούλιο κατάφερε να συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα που έγινε δεκτό από το Ηνωμένο Βασίλειο και ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί μια λύση για εντός αυτού του χρονοδιαγράμματος. Α αφήσουμε όμω τη Μεγάλη Βρετανία στους Βρετανού. Εγώ προβληματίζομαι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτήν ανησυχώ. Τα κακά μαντάτα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να συνεχίζει να ασκεί την ίδια πολιτική της αποτροπής που συνίσταται από δύο σημεία. Πρώτον, της τιμωρίας προς το Ηνωμένο Βασίλειο με, μια έλλειψη συμφωνίας ώστε κανένα στο μέλλον, καμία χώρα στο μέλλον να μην τολμήσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερο στοιχείο αποτροπής είναι η ταπείνωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Παροτρύνοντας τη χώρα αυτή να ακυρώσει το Brexit, οργανώνοντας για παράδειγμα ένα νέο δημοψήφισμα και με το επιχείρημα ότι ήταν οριακή διαφορά, μικρή πλειοψηφία αποφάσισε για την απόσχηση. Αν όμως ήταν το αντίστροφο και είχε συμβεί το αντίστροφο, δηλαδή είχε κερδίσει η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάλι οριακή διαφορά, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θεωρούσε απερίφραστα το αποτέλεσμα δεσμευτικό και μη ανατρέψιμο. Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι η οργάνωση δημοψηφίσματος ε, γίνεται μέχρι ότου λάβει κανείς το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Αυτό είναι η περίεργη συμβολή, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θεωρία και πρακτική της δημοκρατίας. Άλλα κακά μαντάτα είναι αυτή η φοβερή αυταρέσκεια που ακούσαμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα για αυταρέσκεια, αλλά για αυτοκριτική. Ε, πρόεδρε Γιούνκερ και πρόεδρε Τούσκ, ας το παραδεχτούμε. Είχαμε την περίοδο με τις περισσότερες κρίσεις στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και το Brexit είναι μία από τις πολυάριθμες κρίσεις. Και όλοι εσείς που λάβατε ε, τις σημαντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είστε συνυπεύθυνοι και μην αυταπατάστε. Έχετε μεγάλο μερίδιο της ευθύνης και εσείς, κύριοι και κυρίες επίσης. Ο πρόεδρος Μακρόν πρόσφατα έστειλε μια ανοιχτή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρότεινε μεγαλύτερη συγκέντρωση. Και το αστείο είναι ότι χαρακτήρισε αυτή την πρότασή του Ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Μάλλον δεν καταλαβαίνει το νόημα των όρων που χρησιμοποιεί. Καλύτερα Ευρωπαϊκό Λυκόφω θα ήταν πιο δόκιμη έκφραση από το Ευρωπαϊκή Αναγέννηση που χρησιμοποίησε ο πρόεδρο Μακρόν. Σίγουρα το ρολόι του Brexit χτυπά και έχουμε όλη επίγνωση αυτού του γεγονότο. Περιμένουμε πρόοδο από το Λονδίνο, ελπίζουμε να συντελεστεί, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε έκβαση και να είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε ό,τι βοήθεια μπορούμε. Γιατί αυτό θα είναι και δικό μας πρόβλημα, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είμαστε φιλικοί προς οποιαδήποτε απόφαση του Βρετανικού λαού. Πάντως το ρολόι χτυπά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να αφογκραστείτε τους ψηφοφόρους στην Ευρώπη, γιατί όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι ζητούν απεγνωσμένα την αλλαγή και η αλλαγή θα λάβει η χώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φερχόφστατ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να πω στον κύριο Λεγκούτκο ότι είναι λάθος αυτό που ανέφερε, ότι υπάρχει αίσθηση ή επιθυμία ταπείνωσης ε, του, ε, της Μεγάλης Βρετανίας. Κάνετε λάθος. Εμείς έχουμε μεγάλο σεβασμό για ένα μεγάλο Κράτο όπω είναι η Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της ε, τιμωρίας ε, και τη ταπείνωσης είναι πρόβλημα των συντηρητικών, των τόρις. Αυτή είναι η ταπείνωση του Βρετανικού λογίου. δέστε λοιπόν την ομάδα σα. ούτε καν ήρθαν, δεν μα έκαναν καν την τιμή να έρθουν. Ο μόνο που είναι εδώ είναι ο κ. Φαρά. και αυτό με εκπλήσει γιατί είχατε εντύπωση ότι θα ήταν κάπου σε κάποια παρέλαση στη Μεγάλη Βρετανία και τώρα βρίσκεται εδώ. μου θυμίζεται όλο και περισσότερο τον ε, Field Marshal Blackadder, ο οποίος ε, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καθόταν στο γραφείο του στο Λονδίνο και εσείς βρισκόσαστε εδώ στο Στρασβούργο ενώ οι δικοί σας οι άνθρωποι ε, κάνουν διαδηλώσεις στο κρύο, στη βροχή. Να λοιπόν πώς και εσείς αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω αυτά που είπε ο Τσότσιλ, ο οποίος είπε και επιτρέψτε μου να παραθέσω, η επιτυχία είναι η ικανότητα να περνάει κανείς από τη μία αποτυχία στην άλλη, χωρίς όμως να χάνεται ο ενθουσιασμός τέλος της παράθεσης. Νομίζω ότι αυτά είναι τα λόγια του Τσότσιλ, τα οποία ισχύουν απόλυτα και σήμερα στη Βρετανική πολιτική, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ισχύουν και για την κυρία Μέη, γιατί σήμερα το απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αν το επιτρέψει ο πρόεδρος Βουλής, γιατί αυτό είναι το σύστημά τους, θα υπάρξουν 16 επιλογές επιτάπητος ε, για, το, για την έξοδο της ε, Μεγάλη Βρετανίας. Άρα δηλαδή βλέπετε δεν έχει χαθεί ο ενθουσιασμός όπως ακριβώς ε, το ανέφερε και ο Τσόρτσιλ με τα δικά του λόγια. Όμως για να είμαστε πιο σοβαροί μετά όλες αυτές τις καταψηφίσεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας, κατά της μη συμφωνίας, κατά του δεύτερου δημοψηφίσματος, ενδεικτικά τα λέω, ίσως τελικά στο τέλος του τούνελ να φαίνεται λίγο φως διότι με την έγκριση της τελευταίας τροπολογίας για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεων ενδεχομένως να υπάρξει κάποια λύση η οποία θα βασίζεται στην διακομματική συνεργασία, συνεργασία ανάμεσα στους εργατικούς και τους συντηρητικούς. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τίθεται ένα υπαρξιακό θέμα όπως είναι το Brexit και αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με διακομματική συμφωνία στο ίδιο το Κοινοβουλίο. Όπως κάνουμε και εμείς εδώ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, το να τους δώσουμε χρόνο μέχρι τις 11 Απριλίου αυτό θα βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να διαλέξουν ανάμεσα ε, στο να παραμείνουν, στο να υπάρξει μια ε, συμφωνία με κάποια λογική. Γιατί όλοι αυτοί που τα στηρίζουν αυτά πρέπει να συμφωνήσουν. Εγώ δεν υπολογίζω αυτούς που είναι σκληροί με το Brexit γιατί αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τη χώρα. Αυτοί ενδιαφέρονται για την τη δύναμη πώς θα διαμορφωθεί αυτή ε, μέσα στο συντηρητικό κόμμα. Και νομίζω το έχω πει, θα το επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι εμεί είμαστε ανοιχτοί να υπάρξει αυτή η συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία, να ε, υπάρξει μια πολιτική δήλωση με την εξή έννοια. Πρώτα απ' όλα, οι ε, εξελίξεις και η δήλωση να είναι πιο δεσμευτική και για τι ε, δύο αντισυμβαλόμενα μέρη και δεύτερον να μπορούμε μέσα σε αυτήν την πολιτική δήλωση να προβλέψουμε πιο ουσιαστικέ σχέσει ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο από ό,τι προβλέπεται μέχρι τώρα σε οποιαδήποτε πολιτική δήλωση έχει υπάρξει. Και για να τοποθετηθώ και στην τελευταία σα παρέμβαση κύριε Τούσκ θεωρώ ότι Όχι τώρα, δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ω εσεί. Γενικά είμαι αισιόδοξο, αλλά όχι τόσο εσεί. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όχι τώρα, αλλά μετά από κάποιε γενιέ η Μεγάλη Βρετανία θα επανέλθει. Θα επανέλθει στην οικογένεια των Ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί εκείνη η θέση τη, εκείνη η θέση τη Μεγάλη Βρετανία, να είναι μέσα και όχι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω ε, δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει αργότερα και η θέση της Μεγάλης Βρετανίας υπάρχει. Μην ξεχνάμε το 1 εκατομμύριο Βρετανούς που διαδήλωσαν στο Λονδίνο, ε, τα 6 εκατομμύρια υπογραφών και τέλος όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών Κύριε Μπαρνιέ και κύριε Γιούγκερ, γνωρίζω ότι υπάρχει μονόπλευρη και μονομερής ε, δέσμευση της Μεγάλης Βρετανίας για το σεβασμό των πολιτών και εσείς ε, προς τον κύριο Μπάρκλεϊ δεσμευτήκατε ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο και για τους Βρετανούς που ζουν εδώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον έχει έρθει η στιγμή να συζητήσετε με τον κύριο Μπάρκλεϊ και με τα κοινοβούλια για να βρείτε μία λύση πώς μπορούν αυτά να θεσμοθούν νομοθετηθούν έτσι ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν συμβεί και το πιο ανόητο, δηλαδή αν δεν υπάρξει συμφωνία, τουλάχιστον οι πολίτες να μην γίνουν θύματα αυτή της διελκυστίνδα που βλέπουμε να, ε, να διαμφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος, η κυρία Σμιθ έχει το λόγο. Ο κύριος Σμιθ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, τι τραγωδία είναι το Brexit. Υπάρχουν τόσα θέματα που πρέπει να τα δούμε όλοι μαζί και ε, δεν γίνονται λόγω μιας καταστροφής που μόνοι προκαλέσαμε. Ακόμη δεν έχει αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο τι ακριβώς θέλει. Ακόμα δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει ομοφωνία. Γίνεται ε, ε, προσπάθεια να αποκρισταλωθεί μια θέση. Ε, υπάρχουν πολλοί που θέλουν την ανάκληση του άρθρου 50. Κάθε κόμμα στη Σκοτία ε, συμφωνεί ότι το καλύτερο Brexit είναι το μη Brexit. Παρακαλώ συνάδελφοι, μην κλείσετε τις πόρτες σε μας. Πολλοί εργάζονται σκληρά για να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση, να, να υπηρετήσουν τους πολίτες μετά από 15 χρόνια μπορεί να είναι ε, ε, ε, η τελευταία μου αγόρευση. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με την αύξηση του λαϊκισμού. Δεν γνωρίζομαι. Γνωρίζω όμως την Σκοτία ως ευρωπαϊκό έθνος. Ορτάζομαι τη διεθνή αλληλεγγύη, την ελευθερία διακίνησης. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εφεύρουμε κάτι παρόμοιο και η Σκωτία θα ήθελε να ανήκει σε αυτό. Εσείς ε, ως ειδικοί θα πρέπει να ε, σεβαστείτε το Σύνταγμα, θα σεβαστείτε τους ε, συνομιλητές, ε, το, το, το, σέβομαι αυτό. Αν η σκοτία όμως απομακρυνθεί ενάντια στη θέλησή της από την ε, ε, ε, ευρωπαϊκή οικογένεια, αν απομακρυνθούμε ενάντια στη βούλησή μας, η ανεξαρτησία θα είναι η μόνη λύση. Ε, δεν θέλω να υψέλθετε στις εσωτερικές μας συζητήσεις. Αφήστε όμως ένα φως να καίει για να μπορούμε να βρούμε το δρόμο να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Ευχαριστώ. Για την Ενωμένη Αριστερά, εκ μέρου Ενωμένη Αριστερά, ε, το λόγο έχει η κυρία Τσίμα. Κύριοι Πρόεδροι, Βασικά, ε, εδώ και αρκετό καιρό έχουμε κουραστεί να ακούμε συνέχεια τι ίδιε συζητήσει, ε, να μην λαμβάνουμε καμία συγκεκριμένη απάντηση για το τι θα γίνει τελικά. Και μπροστά σε αυτό το δίλημα που προκλήθηκε για διάφορους λόγους, ε, δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από αυτό το δίλημα. Και πρέπει να επισημάνω ότι εμείς ε, νιώθουμε απόλυτο σεβασμό για τους ανθρώπους ε, που σε ένα δημοψήφισμα αποφάσισαν θέλουν να αποχωρήσουν. Σεβόμεθα απόλυτα τους ανθρώπους εκείνους που το τελευταίο Σαββατοκύριακο διαδήλωσαν στο Λονδίνο. Σεβόμεθα απόλυτα όλους εκείνους που υπέγραψαν στο διαδίκτυο ε, το αίτημά τους και νιώθουμε απόλυτο σεβασμό για εκείνους που στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγούν, θα φυγούν απεριόριστα από το Brexit. Νιώθουμε απόλυτο σεβασμό και στον, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επίκυνται οι ευρωεκλογές. Γνωρίζουμε ότι ε, μπορούν οι ψηφοφόροι να στείλουν τους εκπροσώπους τους εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, αυτό όμως ε, θα έχει νόημα για τους ψηφοφόρους όταν οι εκπρόσωποι τους θα είναι εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχει νόημα να έρθουν για έξι μήνες. Σεβόμαστε απόλυτα τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν επιτέλους να ακούσουν μια απάντηση. Κύριε Τούσκα, κύριε Γιούγκερ, σας παρακαλώ πολύ να ασχοληθείτε περισσότερο με τη συζήτηση για τα δικαιώματα των πολιτών, οι οποίοι την ημέρα μετά το άτακτο Brexit θα είναι πολίτες τρίτων κρατών. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δική τους τη ζωή, τη δική τους την ασφάλεια, τους ε, ε, συγγενείς τους, τις οικογένειές τους και λέω λοιπόν και το υπογραμμίζω αυτό συνειδητά, απευθυνόμενοι στην Ιρλανδία, στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και στη Βόρεια Ιρλανδία, ότι ακόμα και αν δεν υπάρξει κάποια λύση σχετικά με την έξοδο από την Τελωνιακή Ένωση, από ε, την κοινή αγορά, θα πρέπει να ισχύει η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Να μην υπάρξει σκληρό σύνορο. Και το λέω αυτό σεβόμενοι απόλυτα τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας στην Ιρλανδία. Εάν λοιπόν θελήσουν να υπάρξει ένα δημοψήφισμα για την ενότητα της δικής τους της νήσου, εμείς τουλάχιστον θα τους στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου ε, της ομάδα άμεσης ε, ελευθερίας, ο κύριος Φάρατ. Ω πρώην Πρωθυπουργό, θα γνωρίζετε ότι ο Μάρσελ Χέικ το 1040 ε, έσωσε από την ε, γερμανική κατοχή μια ε, βελγική πόλη. Και επίσης και στο δυτικό μέτωπο ήταν η Μεγάλη Νίκη της Βρετανίας. Οπότε κανονικά θα έπρεπε για εσάς τους Βέλγους να είναι ήρωας αυτός ο στρατηγός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνέβη στην, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν μια εθνική ταπείνωση και ένα διέξοδο. Γιατί έχουμε την κυρία Τερέζα Μέη, μια πρωθυπουργό που δεν έχει το θάρρο, δεν έχει το όραμα, να τηρήσει τις επανειλημμένες της υποσχέσεις. Να μας βγάλει δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Μαρτίου, αυτή την Παρασκευή. Αυτό δεν συμβαίνει. Και γινόμαστε μάρτυρες ε, Μία ε, προδοσία σε αργή κίνηση, τη μεγαλύτερη ίσω προδοσία στην ιστορία του έθνου μα. Και ο λόγο είναι αυτή η συμφωνία περί αποχώρησης, συνθήκη περί αποχώρησης. Και ε, επιστρέφω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κερδίσαμε τον πόλεμο, αλλά έχουμε τη συνθήκη ε, των Βαρσαλιών, που έχουμε το σύγχρονό τη ισοδύναμο αυτή την συνθήκη, τα 35 δισεκατομμύρια που πρέπει να πληρώσουμε και δεν παίρνουμε σαν αντάλλαγμα τίποτα. Έχουμε την προσάρτηση ενό τμήματο τη εθνική μα επικράτεια με τη μορφή τη Βόρεια Ιρλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ κακή αυτή η συνθήκη, είναι απαράδεκτη, δεν είναι Brexit και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εγκριθεί. Ξέρω ότι όλοι έχετε ε, ε συναρπαστεί και περιμένετε εναγωνίες τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και αν θα διαλέξει κάτι μεταξύ τη Ελεύθερη Διακίνηση και τη Ελληνική Ένωση μια συμφωνία. Αλλά ακόμη και αν το κάνει ε, η Βουλή, κάτι που είναι αναπόφευκτο είναι ε, η παράταση του άρθρου 50. Και θα πρέπει να διαρωτηθείτε, θέλετε όντως μια παράταση του άρθρου 50, θέλετε όντως το Brexit να κυριαρχεί την επόμενη διετία στα προγράμματα εργασιών σας, αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες φιλοδοξίες σας. Θέλετε όντως το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στις τελευταίες ευρωεκλογέ και να στείλει πολλούς ε, ευρωβουλευτές που θα είναι θειασότες της απόσχησης ε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει ακόμη υποστήριξη. Θέλετε να επιστρέψω κι εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε σίγουροι. Ορίστε. Και όλα αυτά προς τι. Το Brexit ούτως ή άλλως θα λάβει χώρα. Κύριε Τούσκ, αν λέτε ότι έχουν ε, αλλάξει γνώμη οι Βρετανοί, ε, απατάστε. Γιατί δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε 15 με 20% διαφορά ε, υπέρ του, της αποχώρησης. Και μάλιστα και νέο δημοψήφισμα να γίνει πάλι η αποχώρηση θα κερδίσει. Ε, κύριε Γιούγκερ ε, Μπαρνέ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς προετοιμαστήκατε για το σενάριο της μη ε, συμφωνίας. Και αυτό δείχνει μεγάλο επαγγελματισμό. Δείχνει ότι ακόμη και αν αποχωρήσει χωρίς συμφωνία δεν πρόκειται να σημειωθούν φοβερές διαταραχές. Ούτε θα διαταραχθεί υπερβολικά η Βόρεια Ιρλανδία. Θα ήθελα λοιπόν να πω προς όλους τους εθνικούς ηγέτες ότι θα πρέπει να απορρίψετε την παράταση πέραν της 12ης Απριλίου. Αφήστε το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει και να συνεχίσουμε όλοι επιτέλους τη ζωή μας. Ο κύριος Ποτέ πριν ε, στην ιστορία, τη μακραίωνα ιστορία της Βρετανίας ε, δεν αντιμετωπίσαμε τέτοια μεγάλη ταπείνωση. Ποτέ πριν δεν κυβερνήθηκαν οι Βρετανοί από συνεργάτες, κουίσλινγκς, προδότες με τρόπο χωρίς προηγούμενο ε, μια νίκη μας αφαιρέθηκε και έχουμε τώρα μια συμφωνία παράδοσης μπροστά μας. Ποτέ δεν μας είχε νικήσει μια ξένη δύναμη. Εκείνη που ε, προάσπιζαν την ε, ελευθερία μας την θυσίασαν ε, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα η τελική παράδοση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακόμα πρέπει να παρακαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν φύγει η Βρετανία στις 29 Μαρτίου, αυτό θα είναι το επίσημο τέλος της δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κανένας λαός που επιθυμεί να είναι ελεύθερος δεν μπορεί να είναι, παραμένει δούλος για πάντα. Η συμφωνία αποχώρησης, οι συμφωνίες για μελλοντικέ σχέσεις, καμία συμφωνία δεν μπορεί να ε, εγκλωβίσει ανθρώπους που δεν θέλουν δεσμά. Μπορεί να ανακληθεί μια συμφωνία στο κοινοβούλιο. Κανένα κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεσμεύσει ένα μελλοντικό κοινοβούλιο. Το Βρετανικό Σύνταγμα θα αποδειχθεί ισχυρότερο, πιο ανθεκτικό από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή συμφωνία ή συνθήκη. Μπορούμε ακόμα να φύγουμε στις 29 με τη χάρη του Θεού. Αν δεν φύγουμε όμως τότε το κόμμα της ανεξαρτησίας της Βρετανίας θα οδηγήσει τον αγώνα για να απελευθερώσει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια και αν χρειαστεί θα αρχίσουμε στις επόμενες ευρωεκλογές το Μάιο. Κυρία ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Παρασκευή 29 Μαρτίου θα έπρεπε να είναι ιστορική ημέρα, μεγάλη σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια μέρα όπου μετά από 40 χρόνια ένταξη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ηνωμένο Βασίλειο πάλι θα είναι ανεξάρτητο έθνος. Ένα έθνος κράτος που θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά απαλλαγμένο από το θεματολόγιο των Βρυξελών. Ε, χωρίς έλεγχο ε, της μοίρας του. Μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεις η Πρωθυπουργό ε, προχώρησε σε ένα σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που υπέβαλε στη Συνεβουλή των Κοινοτήτων. Η Βόρεια Ιρλανδία θα έπρεπε να φύγει με διαφορετικούς όρους σύμφωνα με τον backstop. Συμφωνία για την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας λέει ότι δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα αποχώρησης. Ε, θέλουμε να ε, φύγουμε με συντεταγμένο τρόπο, αλλά η συμφωνία αυτή θα υπονομεύσει την συνταγματική και οικονομική ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι τίμημα που εμείς ε, ε ως ενωτικοί ε, είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε. Τέλος, μια συμβουλή προς, τον, προς τους κυρίους τους και Μπούλμαν. 17,4 εκατομμύρια Βρετανοί ψηφοφόροι είπαν ότι είναι υπέρ της αποχώρησης. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι δημοκρατικές τους επιλογές. Μην κατηγορούμε άλλους. Κύριε Φερχόφστα, το Βρετανικό Κοινοβούλιο ήδη εψήφισε υπέρ μονόπλευρης συμφωνίας γύρω από τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, θα πρέπει να προχωρήσει και στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Η συμφωνία του Μπέλφαστ ε, ε, βασίζεται στην αρχή της συνένεσης. Μόνο με τη συνένεση του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας, κυρία Τσίμερ, θα γίνουν οποιασδήποτε κινήσεις προς αλλαγή του συνταγματικού καθεστώτος της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλά θα κάνετε να το θυμάστε αυτό. Ο κύριος Λεβαντόφσκι έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα πρέπει ε, στη, στην πατρίδα μου να εντυπωσιαστούν από τα λόγια του κ. Λαγκούτκο που έδειξε συμπάθεια προς τη Μεγάλη Βρετανία και προς την έξοδο. Κι όμως ε, ε μπορεί ο κ. Λαγκούτκο να θέλει έξοδο και της Πολωνίας, αποχώρηση της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μη κελιάτε. Το μάθημα και το πάθημα του Brexit θα πρέπει να το θυμηθούμε και στην Πολωνία και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Ο το μόνο αποτέλεσμα, το μόνο θετικό αποτέλεσμα του Brexit είναι οι μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης ε, η σιωπή εκείνων που ε, από το 2016 ε, προαλήφονταν ως διάδοχοι του Brexit. Τελικά η ιστορία του Brexit μας δείχνει τα ιστορικά αποτελέσματα της ανευθυνότητας όταν βάζουμε μια κοινωνία μπροστά σε μια υπαρξιακή επιλογή και δεν ε, δίνουμε μια λύση για τη συνέχεια μετά από την επιλογή και τις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια επιλογή για την κοινωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γουαλτιέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο μέρες μας χωρίζουν μόνο από την ημερομηνία που κανονικά θα έπρεπε να λάβει η χώρα το Brexit. Και ακόμη δεν γνωρίζουμε πότε, πώς, ακόμη και αν τελικά θα συντελεστεί το Brexit. Αυτά, ε, αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγει αυτή η διαδικασία η Βρετανική κυβέρνηση. Αλλά επίσης λέει πολλά για τα ψέματα και τις φαντασιώσεις που έσπηραν εν ώψη του Brexit και πριν το δημοψήφισμα οι θειασότες του Brexit. Τώρα όλα αυτά καταραίουν μπροστά στην πραγματικότητα και τα ανταλλάγματα που θα έπρεπε να δώσει για την κατάσταση αυτή. Και όλη αυτή η πραγματικότητα πια είναι ξεκάθαρη στα μάτια των εκατομμυρίων Βρετανών πολιτών που κατέβηκαν στους δρόμους, κάνουν συλλαλητήρια ζητώντας ένα νέο δημοψήφισμα και ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα τους. Είναι επίσης σαφές ότι η λύση για το αδιέξοδο θα βρεθεί στο Λονδίνο, όχι εδώ στο Στρασβούργο ούτε στις Βρυξέλλες. Η ψηφοφορία της Δευτέρας ε, στην Βουλή των Κοινοτήτων έδωσε μία γραμμή ίσως διεξόδου από αυτό το αδιέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να ε, δει τι θα κάνει με τον έλεγχο που ανέκτησε τις διαδικασίες του Brexit. Επίσης είπαμε ότι η πολιτική διαδήλωση, η πολιτική διακήρυξη μπορεί να αναθεωρηθεί για να χαράξει το δρόμο για στενότερη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα, αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι δυνατό. Αντίθετα, αν η Βουλή των Κοινοτήτων δεν ε, καταλήξει σε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της Τελωνιακής Ένωσης, της ενιαίας αγοράς ή δεν υιοθετήσει την συγκεκριμένη συμφωνία, τότε θα πρέπει να κάνει κάποιες σοβαρές επιλογές. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να ζητήσει πιο μακροπρόθεσμη παράταση, φυσικά αυτό δεν θα γίνει για αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας περί αποχώρησης. Αυτή έχει κλείσει, έχει κλειδώσει και δεν μπορεί να υποβληθεί και πάλι σε διαπραγματεύσεις. Αν όμως το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσει παράταση για να ξανασκεφτεί το Brexit για να ζητήσει στενότερε σχέσει ή να διοργανώσει εκλογέ ή δημοψήφισμα, τότε θα στηρίξουμε το ψήφισμα για μεγαλύτερη παράταση. Ο πρόεδρο τους και ήταν ανέκαθεν σαφέστατο. και το είπαμε και στην ομάδα μας. Έχουμε την αίσθηση τη ε, ε, ιστορικής σημασίας αυτής της κατάστασης. Είχαμε ανέκαθεν ε, επαναλάβει ότι σεβόμαστε το ε, δημοψήφισμα, αλλά να αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να μην φύγει, θα το γιορτάσουμε και δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα για να αποτρέψουμε μια τέτοια πιθανότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπα στην αρχή ότι ε, θα ξεπεράσουμε αυτή την ημερομηνία και δεν έχω απογοητευτεί. Είχα πει ήδη από την αρχή ότι ο λαός που εγώ εκπροσωπώ ποτέ δεν θα δεχθεί ε, ένα σύνορο ε, στην ε, Ιρλανδική θάλασσα. Γι' αυτό ακόμη υπάρχει, κύριε Μπαρνιέ, κύριε Γιουνκέρ. Επίσης, το backstop για την Ιρλανδία και μια ακύρωση μιας διεθνούς συμφωνίας, για τις συμφωνίες του Belfast, θα δημιουργήσει μια πολύ αρνητική κατάσταση. θα πρέπει να αγνοούμε το πνεύμα εκείνη τη συμφωνία. Επίση θα πρέπει να ακούσουμε του πάντε στη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι μόνο εκείνου που ε, ε, φωνάζουν πιο δυνατά. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία στη Βόρεια Ιρλανδία που θέλει ένα καλό δρόμο, μια καλή λύση για τη Βόρεια Ιρλανδία, για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις θέσεις του παρελθόντος και να αναζητήσουμε ένα καλύτερο μέλλον στο οποίο θα μπορούσαμε όλοι να συνεργαστούμε. Εξακολουθώ να προβληματίζομαι και να έχω ανησυχίες ότι διατρέχουμε και πάλι τον κίνδυνο να συγκρουστούμε με τείχο. Όχι επειδή φταίει ο κύριος Τούσκο, ο κύριος Μπαρνιέ ή οποιοδήποτε άλλος. Υπάρχει όμως κίνδυνος να αποτύχουμε και ελπίζω να φροντίσετε να αποτρέψουμε μια τέτοια σύγκρουση με τον τείχο. Και επίσης θα μπορούσαμε όπω είπε ο συνάδελφο από τη Σκωτία, να είναι και ο δικό μου τελευταίο λόγο μετά από μία τριακονταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πολύ καιρό, το απόλαυσα και έχω πολύ θετικέ ενημνήσει. Ελπίζω να ε, εκπροσώπησε επάξια το λαό της Βορειοορλανδίας. Ευχαριστώ. Mr. Nicholson, how thoughtless of me. Κύριε Νίκολσον, ε, λάθος, λάθος ε, εκ μέρους μου το να μην σας σεβαστώ